διαμαρτυρίας ε, κατά της μονομερούς επιβολής των συνδικών εργασία από την διοίκηση και ε, δυστυχώ πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η διερμή θα σταματήσει την ώρα που προβλέπεται η λήξη της συνεδρίας. Ευχαριστούμε. Okay. <clears throat> We begin by item 9. Αρχίζουμε, λέει ο πρόεδρο. Είμαστε στο σημείο υπαριθμών 9, που είναι οι ανακοινώσει του Πρόεδρου. Να σας διαβάσω τώρα τις αποφάσεις των συντονιστών. Πρόκειται για μακρύ κατάλογο αυτών. Οπότε έχουμε και λέμε. Χθες στη συνάντησή τους, το χθες το απόγευμα, απεφάσισαν το εξής. Κυρία Φεράρα, πρόκειται να οριστεί ως ε, εισηγήτρια για την άρση ασυλίας του κυρίου Γεωργίου Κίρτσου και του κυρίου Σιβιεύκα. για τον κύριο Μπριουά και την Σοφή Μόντελ. Ο κύριος Σβιεύκα θα είναι ο εισηγητής για την έκθεση των ψηφιακών εργαλείων και μηχανισμών όσον αφορά το εταιρικό δίκαιο. ΔΕΜΕΚ. Ο εισηγητής για το άρθρο 54 γνωμοδότηση της ΣΥΜΚΟ όσον αφορά την διαφάνεια για τις επιχειρηματίες όσον αφορά τις ε, Ιντερνετικές υπηρεσίες δημοσιολάβησης. Μπερζερό, συγητής για την ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και όσον αφορά και την εφαρμογή ε, της σχετικής διάταξης. Χάουδαλα η για τη γνωμοδότηση όσον αφορά τις ε, υποχρεώσεις για την ευθυγράμμιση περιβαλλοντικής πολιτικής Ντελβό. Η συγγήτρια για την γνωμοδότηση για τη μείωση των επιπτώσεων κάποιων πλαστικών προϊόντων επί του περιβάλλοντος. Η κυρία Γκέμπαρτ, η συγγήτρια της γνωμοδότησης για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη 2021 έως 2027. Ο κύριος Λεμπρετό γνωμοδότηση για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 και η κυρία Κάουφμαν για την γνωμοδότηση του προγράμματος για αξίες και δικαιώματα. Αποφασίσαμε να μην γνωμοδοτήσουμε όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα. Επίσης αποφασίστηκε το εξής. να γνωμοδοτήσουμε όπως μας ζητήθηκε προς την ΑΒΚΟ με τη μορφή επιστολής όσον αφορά την κατάσταση της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης και ο υποφαινόμενος πρόκειται να είναι ο εισηγητής. Να μην γνωμοδοτήσουμε όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και την προστασία της εξοδαφικής εφαρμογής της νομοθεσίας τρίτης χώρας. Να γίνει ακρόση για την πρόταση της ε, συλλογικής αποκατάστασης βλάβης και επίση ε, για την στρογγυλή τραπέζα όσον αφορά την επιλογή ανωτέρων υπαλλήλων, ανωτέρων στελεχών, σύμφωνα με την πρακτική, την πάγια θα έχουμε πρόεδρο ε, και θα δοθεί εντολή σήμερα από την Επιτροπή όσον αφορά τις τροπολογίες του προϋπολογισμού του 10. Να περιμένουμε επίσης να ψηφίσει η ΙΜΚΟ πριν γνωμοδοτήσουμε για τις νομικές βάσεις της πρότασης ΣΜΙΤ. Να αναλάβουν πρωτοβουλία διαβίβασης επιστολής όσον αφορά ε, την πρόσληψη προσωπικού για την γραμματεία μας. Για την εβδομάδα 26 απεφάσισαν οι συντονιστές πρώτον να ορίσουν τους εξής μόνιμους συζητητές για την περίοδο μισό λεπτό συμπαθάτε με. Επαναλαμβάνω, ο Πρόεδρος. Οι ακόλουθοι μόνιμοι ζήτητες για την περίοδο 1η Εβδόμου έως 31η Δωδεκάτου ου έτος και ως για τις νομικές βάσεις ο κύριος Λεμπρετών για επικουρικότητα Φεράρα για τις διαφορές Χάουταλα για την ε, προσωπία των ε, πράξεων, Γκάγκα, ως εισήδρια για ε, επαναδιατύπωση και κωδικοποίηση ή κωδικοποίηση και επαναδιατύπωση. Επίσης, αποφασίστηκε στις 27 Νοεμβρίου του 2018 να έχουμε μια διακοινοβουλευτική συνάντηση με την ΠΕΤΗ όσον αφορά την χειραφέτηση των κοινοβουλίων για το κοινωτικό δίκαιο. Επίσης, να συνεχθούμε με τον συντονιστή του ΕΛΚΟ να αυτά τα δικαιώματα των ανηλίκων για τις διαφορές διασυνοριακών οικογενειών και επίσης ότι πρόκειται έτσι να περιφερθούν τα δικαιώματα των ανηλίκων ε, τον Νοέμβριο του 2018 το απόγευμα κάποια μέρα, οπότε θα, θα έχει χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αναβάλουμε την ακρόαση όσον αφορά την ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη για μετά την αποστολή ή στο Μομπελιέ και θα οριστεί κάποια στιγμή η συγκεκριμένη ημερομηνία. Τελευταίο είναι το να ε, γίνει μία ακρόαση όσον αφορά την ταχεία διαδικασία για το θέμα που συζητήσαμε χθε όσον αφορά τι εμπορικέ διαφορέ. Επίση, συμφωνήθηκε σήμερα το απόγευμα οι πλαστικές φιάλες με το νερό που συνήθως μοιράζονται στην αίθουσα να αφαιθούν και να διαθέσουμε στην είσοδο της αίθουσας. Αυτά και συνεχίζουμε. Και πάμε στο σημείο παρθεμών 10 ανταλλαγή απόψε αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές. Κύριε έχετε το λόγο, συγητής. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόσφατα ορίστηκα εισηγητή στη γνωμοδότηση που θα καταρτήσει η Επιτροπή μας για, την, ε, για τα αυτόνομα οχήματα. Δυστυχώς, Κατά την προετοιμασία της γνωμοδότησης ε, βρεθήκαμε υπό μεγάλη πίεση λόγω των ε, προθεσμιών που έθεσε η Επιτροπή Μεταφορών που είναι και η καθέληνα αρμόδια έτσι ώστε να μπορέσει να εγκρίνει την έκθεσή της εγκαίρως. Πρέπει αμέσως μετά το καλοκαίρι να έχουμε καταρτήσει την γνωμοδότηση και να ψηφίσουμε το τελικό κείμενο τον Οκτώβριο έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη στην τελική έκθεση την οποία θα ψηφίσει η Επιτροπή Μεταφορών τον Νοέμβριο. Δεν έχουμε λοιπόν πολύ χρόνο και δεδομένου τούτου θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να καλύψει η γνωμοδότηση. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της ε, δικής μας Επιτροπής καλύπτει μόνο την αστική ευθύνη και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα μπορούσε επίση η Επιτροπή μας να είναι αρμόδια για τις πτυχέ ε, που αφορούν νέε τεχνολογίες. Επίσης, η ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από την χρήση των αυτόνομων οχημάτων είναι κάτι που θα μπορούσε να μας αφορά. Δεδομένης της ε, εξέλιξης της τεχνολογίας, θεωρώ πως τόσο η βιομηχανία όσο και οι καταναλωτές χρειάζονται σαφείς πανευρωπαϊκούς κανόνες έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι εξελίξεις και οι καταναλωτές να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο από τους νέους κινδύνους που απορρέουν από την ε, χρήση αυτόνομων οχημάτων, χωρίς οδηγό δηλαδή. Επομένως θα έπρεπε να διευκρινιστεί ποιος είναι ο υπεύθυνος σε περίπτωση ε, ζημιών. Δυστυχώ, όμω δεν έχουμε προχωρήσει τόσο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσεις που έχουν προκύψει από την τεχνολογία των αυτόνομων οχημάτων. Ίσως θα μπορούσαμε να διακρίνουμε κάποιες κατηγορίες κινδύνου, τις οποίες νομίζω θα δούμε και στην πράξη λόγω της πρόοδου της τεχνολογίας. Πρώτον, πρώτη κατηγορία, οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με βλάβες από το λογισμικό λειτουργίας που χρησιμοποιεί το όχημα. Δεύτερη κατηγορία. Κίνδυνοι από βλάβες δικτύου. Τρίτη κατηγορία. Κίνδυνοι που απορρέουν από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Και τέταρτη κατηγορία. Ε, κίνδυνοι και άλλοι εξωτερικοί, εξωτερικοί παράγοντες από τη χρήση διαφόρων προγραμμάτων. Αυτά είναι ελάχιστα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Θα υπάρξουν πολύ περισσότερα και αν δεν βρούμε κατάλληλη λύση θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στα αυτόνομα οχήματα, το οποίο με τη σειρά του θα επιβραδύνει την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την αξία που θα προκύψει προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε λοιπόν αρκετές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, τους περιορισμούς και τις ελλείψεις στο εφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όσον αφορά την ευθύνη των ε, χρηστών και των μερών. Έπειτα. Χρειάζεται να προσαρμόσουμε τους υφιστάμενους κανόνες ή να εισαγάγουμε νέους. Και τρίτον, χρειάζεται να σκεφτούμε νέους ε, δικονομικούς κανόνες όσον αφορά τις ε, ζημίες που προκαλούν τα αυτόνομα οχήματα. Επιπλέον, πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα που θα προκύψουν ε, στον χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά θέματα ρομποτικής και αυτόνομων οχημάτων, όμως οι υφιστάμενοι κανόνες θα μπορούσαν να τροποποιηθούν, να προσαρμοστούν με τη δέουσα προσοχή στη διαδικασία. Επίσης, να μην ξεχνάμε πως πρέπει να υπάρχει μια εξισορροπημένη προσέγγιση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, του υλικού και του λογισμικού, να προστατευτεί η καινοτομία και να, δοθεί ταυτόχρονα, να δοθούν ταυτόχρονα ε, κίνητρα για την προώθησή της. Και τέλος, να αναπτυχθούν διάφορες προϋποθέσεις για ε, την πνευματική ιδιοκτησία, για, ίσως με, τον, με τη μορφή κάποιων ε, τεστ, για αυτά τα αυτόνομα οχήματα και αυτά θα έπρεπε να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την προσοχή σας και θα χαρώ να ε, ανταλλάξουμε απόψεις. ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κάουφμαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, ο κύριος Βόλκεν δεν μπορούσε να έρθει αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό λοιπόν και μου ζήτησε να παρουσιάσω τις δικές του απόψεις. Καλωσορίζουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 17 Μαΐου για μια ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με την κινητικότητα του μέλλοντος και αναγνωρίζουμε το τεράστιο δυναμικό που έχει η αυτόνομη οδήγηση τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα ε, νομικής φύσης τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν. Ε, σε ό,τι αφορά την ευθύνη, σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει καταρχάς να οριστεί σαφώς ποιος έχει την ευθύνη. Είναι ο κατασκευαστής, είναι ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός. Εδώ νομίζω πως είναι απαραίτητη η χρήση και ύπαρξη ενός μαύρου κουτιού το οποίο φυσικά πρέπει να ε, συμφωνεί και με τους ε, κανόνες σχετικά με την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, ε, το θέμα της ευθύνης θα πρέπει να ε, διευκρινιστεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, εκτίμηση του, και τη διαχείριση μάλλον του κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ό,τι αφορά την καταβολή αποζημιώσεων δεν θα, θα πρέπει να διευκρινιστεί επίσης το θέμα της ευθύνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι η οδηγία για την ευθύνη προϊόντων χρειάζεται προσαρμογή για να μπορέσει να συμπεριλάβει και τις νέες τεχνολογίες. Γι' αυτό συστάθηκε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα Γι' αυτό λοιπόν αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα απορίσματα της Επιτροπής αυτής. Σε ό,τι αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, το θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται από το όχημα. Χρειάζεται να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και οι κατασκευαστές των οχημάτων όσο και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις ε, απαιτήσεις και την νομοθεσία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ιδιαίτερα οι ε, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων. Θα πρέπει επίσης να ε, διασφαλίζεται η φορητότητα έτσι ώστε να αποφευχθούν τα διάφορα προβλήματα ε, που οδηγούν σε αποκλεισμό των μικρών επιχειρήσεων από την πρόσβαση στην αγορά. Αυτά έχει να πει ο κύριος Βόλκιν και σας ευχαριστεί πάρα πολύ. Η κυρία Ντελβό έχει στο λόγο. Ναι, θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Ράντερ στα αγγλικά για την παρουσίασή του και συμφωνώ ότι θα πρέπει να περιοριστούμε στις ε, αρμοδιότητες επιτροπής μας, δηλαδή θέματα ευθύνης. Επίσης επισημαίνω ότι υπάρχει μια εξαιρετική έρευνα της EPRS ε, για, την, ε, για τα ζητήματα ευθύνης που προκύπτουν από τα αυτόνομα αυτοκίνητα, όπου επισημάνονται και τα κενά ή τα η ελλείψεις στην νομοθεσία μας σε σχέση με το θέμα αυτό και θα είναι πολύ χρήσιμη πιστεύω στο, στην κατάρτιση γνωμοδότησης. Οπωσδήποτε είναι πολύ απαραίτητη η εμπιστοσύνη στη νέα τεχνολογία. Ιδάλλως ε, δεν θα μπορέσει να απογειωθεί ε, αυτός ο κλάδος και τα αυτόνομα αυτοκίνητα τουλάχιστον θα μπορούν να είναι στους δρόμους, να κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Ε, άρα χρειάζεται αυτή η εμπιστοσύνη. Και δεύτερο, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε σε αρμοδιότητες μας θέματα διεθνούς δικαίου. Φερρυπίνη συστάσεις σχετικές με την ε, σύμβαση της Βιέννης. Γιατί και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή απαιτείται να υπάρχει οδηγός ο οποίος αναλαμβάνει την οδήγηση. Στο μέλλον, πώς θα γίνει η προσαρμογή των υφισταμένων συμβάσεων στη νέα τεχνολογία και τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να κοιτάξουμε μέσα από την έκθεσή μας βέβαια. Άντερσον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Ράντο για την ε, παρουσίαση των προτάσεων. Περιμένω με χαρά να τις διαβάσω. Ο συνάδελφος έχει διαβάσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι την έκθεσή μας για το ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη της Επιτροπής Γιούρι πάντα και χαίρομαι ιδιαίτερος. Ε, ακούω μέσα στις παρατηρήσεις του πολλά από αυτά τα στοιχεία αυτής της εκθέσεως για τα δικαιώματα του πνευματικού δημιουργού. Ε, δημιουργία νέων δικαιωμάτων, νέου τύπου δικαιωμάτων που μπορεί να αντίκεινται στον ελεύθερο ανταγωνισμό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Θα κοιτάξω βέβαια πολύ προσεκτικά τις προτάσεις του ε, συναδέλφου, αλλά πρέπει να προστατεύουμε τον ανταγωνισμό και όχι να τον αποτρέπουμε. Επίσης, Εάν ο σχεδιασμός αυτών των δικαιωμάτων πραγματικού δημιουργού δεν ε, είναι πολιτός ορθός, θα, δράσουν, ε, θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποτροπή ε, του κάθε πνευματικού δημιουργού ή παραγωγού από το να κάνει μια νέα πρόταση, να σχεδιάσει κάτι καινούριο. Θα θυμάστε φαντάζομαι τις προδιαγραφές του Dieselgate όπου δύο ε, σαφώς αυστηρές νομοθεσίες σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία ή την βιομηχανική ιδιοκτησία προκειμένου, δεν επέτρεψε την διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκάλυψη του σκανδάλου ε, στο οποίο ήταν εμπλεκόμενη η Volkswagen με την απόκρυψη στοιχείων εκπομπών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι οτιδήποτε εισάγεται θα επιτρέπει την έρευνα από πλευράς ανεξαρτήτων ερευνητών, επιστημόνων, αυτών των αυτόνομων αυτοκινήτων, ώστε να μπορούν να γνωρίζουν με απόλυτη ασφάλεια οι χρήστε ότι είναι ασφαλή αυτά τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Και εγώ είμαι πεπισμένο ότι θα είναι πολύ πιο ασφαλή από τα αυτοκίνητα που οδηγεί ο άνθρωπο, εφόσον όμω γίνει σωστά, πολύ σωστά ο σχεδιασμό. Και εδώ πέρα ακριβώ είναι όλη η, η σημασία αυτή τη πρόταση. Ο πρόεδρος, περιμένω να αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Προφανώς ο κύριος Άντερσον εγείρει το ζήτημα, το αιώνιο ζήτημα της ε, αντιπαράθεσης ε, δικαιωμάτων πνευματικής διοκτησίας και ε, ανταγωνισμού οπωσδήποτε, χωρί ε, δικαιώματα πραγματική ιδιοκτησία. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανεί να περιμένει ότι θα είχαν αναπτυχθεί τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Κύριο Λεπρετό, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ακούω τον κύριο Ραντεφ και ένα πράγμα έχω να σημειώσω ότι έχει κάνει μια αρκετά διεξοδική εξέταση των κινδύνων σε θέματα τη ασφάλεια. Ιδιαίτερα εμένα με ε, απασχολεί το θέμα της κυβερνοεπίθεσης. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ε, τρομοκρατικό κίνδυνο επί παραδείγματι εξασφάλιση του ελέγχου των αυτόνομων αυτοκινήτων με στόχο να τα χρησιμοποιήσει ο τρομοκράτης για, ε, ως όπλα εναντίον ε, αθών πολιτών. Έτσι λοιπόν ξεπερνούμε τα θέματα και τους κινδύνους, τους κοινού, τα κοινά ζητήματα της αστικής ευθύνης όπως τη γνωρίζουμε πάντα και περνούμε σε άλλα θέματα απειλής και άρα χρειάζεται να έχουμε πάρα πολύ αποτελεσματική προστασία. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ε, κύριε Άντερσον, θέλετε κάτι ακόμη? Ναι, θα ήθελα μόνο να διευκρινίσω ότι εδώ ε, αυτό που είπα δεν είχε στόχο να στραφώ κατά των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αλλά να πω ότι πρέπει καλύτερα να αξιοποιηθούν αυτά που υφίστανται, γιατί δάλλως αν πρόκειται να σχεδιαστούν εξ αρχής, ε, θα είναι πολύ δύσκολο να σχεδιαστούν σωστά. Και φαντάζομαι ο πρόεδρος συμφωνεί με τις προθέσεις μου. Ε, όσο και αν μπορεί να οδείξει σε παρερμηνία η ορολογία που χρησιμοποίησα. Ο πρόεδρος βεβαίως... Ε, νομίζω ότι το ολοκληρώσαμε, εκτός και αν ο κύριος Ράντι θέλει το λόγο, πάλι όχι. Πολύ καλά. Και έτσι αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε προγραμματίσει για τις 10 το πρωί τις ψηφοφορίες μας. Και πάλι λοιπόν ανακαζόμαστε να κάνουμε διάλειμμα για καφέ. Mr. Ο κύριος Μαρίνιου Πίντου. Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή αυτή και από εσάς, κύριε Πρόεδρε, να μας ε, δώσετε μια μετάφραση για τα όσα ελέγχθησαν σχετικά με, την, ε, με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στη χώρα μου έγινε μια μεγάλη συζήτηση, εκτοξεύτηκαν κατηγορίες, ε, υπόθηκαν τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλούμε να ε, μας δώσετε μια μετάφραση, στην περίπτωσή μου στα πορτογαλικά, γιατί Μόνο όταν έχουμε την επίσημη μετάφραση θα μπορέσουμε να κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτά που εγκρίθηκαν. Διαφορετικά υπάρχει παραπληροφόρηση ε, από ορισμένους. Μόνο το αγγλικό κείμενο είναι διαθέσιμο και μάλιστα υπάρχουν κάποια προβληματάκια με τους νομικούς όρους. Ε, σίγουρα βέβαια στα αγγλικά δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όταν όμως ε, μεταφράζεται το κείμενο από την αγγλική ε, γλώσσα σε μια λατινογενή στην περίπτωση αυτή θα υπάρξουν προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να μας δώσετε μια πορτογαλική μετάφραση του κειμένου. So, uh, I'm informed that... Uh, μου λένε... Γίνεται η μετάφραση του εγγράφου. Τώρα το πότε θα τελειώσει, αυτό είναι θέμα της υπηρεσίας μετάφρασης. Ε, βέβαια όμως και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά γιατί είναι ολομέρεια να έχει γίνει μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες εργασίας. το άρθρο 13. Αυτό είδα εγώ. Γιατί στην Πορτογαλία μας κατηγορούν ότι λογοκρίνουμε ό,τι ανεβαίνει στο ίντερνετ. Και ο Γκέμπελς το λέει γι' αυτό. Ψέματα, ψέματα, όλο κάτι θα μείνει. Επομένω να γίνει η μετάφραση του 2013 και να πούμε ότι αυτό εγκρίθηκε και κατόπιν ε, ο καθένας να εξαγάγει τα συμπεράσματά του. Λογοκρισία ή όχι λογοκρισία. Να περιμένουμε, να περιμένουμε τη μεταφραστική υπηρεσία, λέει ο πρόεδρος. Δεν γίνεται η μετάφραση άρθρο-άρθρο. Ε, παραδίδεται μόλις έχει μεταφραστεί όλο το έγγραφο. Διάλειμμα για καφέ μέχρι τις 10, λέει ο Πρόεδρος. So, colleagues, may we begin? Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες και είμαστε στο σημείο 12 της μέρης της διάταξης. Σχέδιο έκθεσης για πρόταση κανονισμού σχετική με το εφαρμοστέο δίκαιο στα αποτελέσματα των εκχωρήσεων με όχι, συγγνώμη, με το ζήτημα του ασύλου. Τροπολογία 5 υπέρ. Αποτελέσματα εκχωρήσεων απαιτήσεων έναν τρίτον. Απεριευθυσυμβαστική πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά επαληθεύουμε τη 41 παρακαλώ I miss my card. Mm -hmm. And what, what was your... It's vote? positive positive. Είπε. Εγκρίνεται λοιπόν. We continue by amendment 6 and 40. Τροπολογία 6 ε, και 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Η 45 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 7 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Από την 8 έως και τη 48 υπέρ. και, μέχρι και 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απεριφθεί. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 65 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 65 So it's 9 to 10. Ε, ναι, λέει ο πρόεδρος, υπέρ 10 κατά, εν απερίφθη. 66 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 68 υπέρ κατά αποχές απερίφθη η 69 έχει αποσυρθεί 16 κατά αποχές εγκρίθηκε 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά απόχες και επαληθεύουμε την 19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 και ψηφίζουμε το σχέδιο πρώτα, στο σύνολό του υπέρ. Όχι ονομαστικά. Ονομαστική ψηφοφορία. Και εγκρίνεται. 17 υπέρ, μία αποχή. Και τώρα την εντολή για τις διαπραγματεύσεις με 13 ψήφους πλειοψηφία παρακαλώ, ονομαστικά. Χρειάζονται 13 ψήφοι για την πλειοψηφία. Δεκαοχτώ υπέρ, ένας, κατά, ένας αποχή και καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια στον ε, υποφαινόμενο και προχωρώ στην πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού 1092-2010 για το η μακροπροληπτική επίβλεψη του χρωματοοικονομικού συστήματος και ξεκινώ με την τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ να επαληθεύσουμε την 9 παρακαλώ απερίφθη. Οχτώ υπέρ, εννέα κατά. Ε, προχωρώ η δέκα και η τρία μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 35 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε την 38. Απερίφθη. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε απερίφθη 12 και 41 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά όχι Για να το επιβεβαιώσουμε λίγο. Ψηφίσαμε την συμβαστική 10, έτσι. Λέει και σας ο καταλογός ότι πρέπει να πάμε στις 47 μετά. Έχει ζητήσει κανείς να ψηφιστεί χωριστά το δεύτερο τμήμα του 14. Κύριος Χρυσόγονος. Ναι, χωριστά. Δεν έπρεπε να είναι στον γκρι. Okay, then it is a mistake. It, it's the mistake in the voting list. Άρα έχει λάθος ο κατάλογος και ψηφίζουμε την τροπολογία 14 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ας το επαληθεύσω. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική παριθμόν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 21 υπέρ, 22, λέει ο πρόεδρος, 22 υπέρ, κατά, να επαληθεύσω την 22. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές επαληθεύουμε την 4 παρακαλώ συμβαστική 4 που δεν φαίνεται να είναι συμβαστική εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σχέδιο γνωμοδότης του συνολό του ηλεκτρονικά And that has been adopted. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Χρυσόγονο. Συνεχίζουμε τώρα με την ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότηση σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 60 αποσύρεται. 59 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 59. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 7 παρακαλώ. That has been adopted. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη 10 παρακαλώ, γιατί δεν είδα πολλά χέρια. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι σίγουρος. Ελέγχουμε λοιπόν. Εγκρίνεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 71. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 και 75 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 78 παρακαλώ. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 79. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 80. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τη συμβιβαστική 7. Εγκρίνεται. 23 και 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 99 υπέρ κατά αποχές Καλύτερα να ελέγξουμε. Την 99. Εκρίνεται. 100. Α, όχι, όχι. Καταπίπτει 100. 101. Ψηφίζουμε ξανά την 99, το ζήτησε η Αντιπρόεδρος. Υπήρξε ένα θέμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 99. Απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στην 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 104. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 27. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 110. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε καλύτερα την 31. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50. Α, με συγχωρείτε, 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό του. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια ξανά στον κύριο Χρυσόγονο. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία για την εντολή προς τον εισηγητή για την κατάθεση τροπολογιών επί του προϋπολογισμού. Σημείο 15. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον υποφαινόμενο. Τελευταία ψηφοφορία. Ενιαία ψηφιακή πύλη ηλεκτρονικά. One more. Μία ακόμα έμεινε. Okay. And that has been adopted. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Φως. So that's all for the votes. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ψηφοφορίες. So, dear colleagues, we continue by items Συνεχίζουμε, συνάδελφοι, με τα 17 και 18. Σημεία της σημείας διάρκειας θα συζητηθούν από εκείνο δυστυχώς. Δεν παρίσταται ο εισηγητής. Αλλά, εκ μέρους του, να σας διαβάσω το σημείωμα το οποίο μας διαβίβασε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως εισηγητής όσον αφορά ε, αυτά τα δύο θέματα θα πρέπει να αναφέρω στην Επιτροπή όσον αφορά τον πρώτο άτυπο τριμερή διάλογο όσον αφορά την ευθυγράμμιση RPS ε, σε συνεργασία με την Προεδρία. Βρίσκεται εν εξελίξη ακόμη ε, επιβουλές Προεδρίας 28 ε, Ιουνίου. Αυτό έγινε ούτως ώστε η εντολή να ξεκαθαριστεί για τα τρία θεσμικά όργανα και να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες σχετικές με τις διαπραγματεύσει. Η εντολή δόθηκε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο από το Συμβούλιο. Οπότε ήρθε η στιγμή να αρχίσουν οι διοργανικές διπραγματεύσεις. Τα τρία θεσμικά όργανα συνεφώνησαν ότι τα πράγματα έχουν οριμάσει αρκετά ούτως ώστε να προχωρήσουμε και το καθεσμικό όργανο παρουσίασε τα στοιχεία της εντολής του πρώτα-πρώτα την αντικατάσταση των κανονιστικών μέτρων με έλεγχο μέσω κατεξοδότηση ή πράξεων ή εφαρμοστικών πράξεων όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά δεύτερο λόγο έχουμε κάποιες πράξεις που εξαιρούνται ή αναστέλλονται, αναβάλλονται. Επίσης να διαγραφεί η εξουδότηση που προβλέπεται σε σχέση με αυτές τις κατηγορίες πράξεις. Επίσης να, να έχουμε αυτό το Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις εφαρμοστικές πράξεις και να γίνει αντικατάσταση από εφαρμοστική σε κατεξοδότηση πράξη για αντιστρόφους. Επίσης να υπάρξει σχετική υποβολή εκθέσεων. Κατά έκτον έχουμε κατεπίγουσα διαδικασία το unbundling και προβλέπεται και προθεσμία ε, υποβολή ένσταση. Να συγχυστεί η δουλειά σε τεχνικό επίπεδο, προτείνει δε το Κοινοβούλιο ότι σε αυτό το τεχνικό επίπεδο θα πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα βασικά στοιχεία της εντολής για τα τρία θεσμικά όργανα. Μπορεί να υπάρξει σύγκληση κατά αυτές τις ε, κόκκινες και κίτρινες περιοχές της ε, εντολής και επομένως θα συνεχιστεί η συζήτηση στο μέλλον σε κάποιον άλλο τριμερή διάλογο. Θα συνεχιστούν επομένως διαπραγματεύσεις επί Αυστριακής Προεδρίας Πρόεδρος Κοινοβουλίου θα πρέπει να σας πω ότι θα είναι επικοδομητικές οι διαπραγματεύσεις και συνεχίζουμε την τεχνική δουλειά με συναντήσεις που θα συνεχιστούν και τον Σεπτέμβριο. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν τον Οκτώβριο σε πολιτικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. So... Αυτά για το 17 και το 18. Συνεχίζουμε τώρα με το 19 και κλεισμένα των θηρών. Οπότε παρακαλώ όλοι οι οποίοι δεν δικαιούνται να παραστούν να αποχωρήσουν.